E, wznawiam posiedzenie. Protokół z wczorajszego posiedzenia jest dostępny wszystkim Państwu. E, chciałem zapytać, czy są jakieś uwagi. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ερωτήσω αν υπάρχουν σχόλια στα χθεσιν, για τα χθεσινά πρακτικά τα οποία σας έχουν διανεμηθεί. Εάν όχι, θεωρώ ότι εγκρίνονται. Σύμφωνα με την ημερήσια κατάσταση, έχουμε δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την κατάσταση των Ρωμά στην Ευρώπη.